Πόσο σημαντική είναι και η Επιτροπή μας. Εμείς πιστεύουμε παρατηρούμε τα γεγονότα, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε τόσο πολλούς θεσμούς Παρόλα αυτά, μεταξύ εθνών υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη μετακίνηση στρατευμάτων Έχουμε και τις εκλογές στη Μολδαβία. Ίσως υπάρχει κάποια σύνδεση Για να δούμε που θα μας οδηγήσουν μήπως σε λίγους μήνες έχουμε πιο δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λυπούμε που δεν μπορώ να μείνω όσο το περισσότερο, αλλά δυστυχώς έχω και εγώ πολύ συχτό πρόγραμμα. Εκτιμώ αυτή την ευκαιρία να μοιραστούμε κάποιες σκέψεις όσον αφορά την κατάσταση προόδου στην Ουκρανία, αλλά και ε, γενικότερα για την ατζέντα του ΟΑΣΕ που έχει αναπτυχθεί με συγκρουσιακό τρόπο θα έλεγα στον οργανισμό. Κάποιες φορές επανέρχομαι στους καιρούς του... της Δασέ και του ψυχρού πολέμου. Εκείνους τους καιρούς θυμάμαι. Είναι μια δύσκολη φάση για αυτόν τον οργανισμό, αλλά γι' αυτό έχει φτιαχτεί αυτός ο οργανισμός για να αποτελέσει μια πλατφόρμα, ένα βήμα συγκέντρωσης, συζήτησης ε, για να προσπαθήσουμε ανάμεσα σε χώρες που έχουν μεταξύ τους δύσκολες ε, σχέσεις να βρούμε έναν κοινό παρονομαστή ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Αυτό που βλέπουμε σήμερα στην Ουκρανία είναι μεγάλη ταχύτητα στην πολιτική διαδικασία και την πολιτική εφαρμογή της ε, συμφωνίας του Μίνσκ. Βλέπουμε να υπάρχει ε, διαρκώς ε, ε, οπισθοδρόμηση, διολίστηση προς τα πίσω. Βλέπουμε ότι οι γραμμές που είχαν οριστεί στη διάρκεια της ανακοχής έχουν κινηθεί, στρατιωτικές αλλαγές έχουν συνεχίσει σε ολόκληρη αυτή τη φάση, έχουν ενταθεί στο τελευταίο καιρό. Είδαμε κονβόι με βαριά όπλα, φορτηγά, πυρομαχικά, τάγκς να μπαίνουν στην περιοχή όπου ίσχυε η ανακοχή, η πάυση του πυρός και βέβαια έτσι ενίσχυση της δυνατότητας ε, στατικών επιχειρήσεων σε αυτήν την περιοχή. Ταυτόχρονα Διαρκή εμπόδια διαπιστώσαμε στην δυνατότητα ε, να ασκήσουμε εμεί τι δικέ μα λειτουργίε, όπω είχαμε συμφωνήσει το Και εμεί έχουμε περιορισμένη πρόσβαση, έχουμε κάποιε ομάδε ε, στο Ντούγκανς και στο Ουνιέτς, αλλά αυτές οι ομάδες έπρεπε να μπορούν να κινηθούν πέρα από αυτές τις ε, τοποθεσίες. Ε, αυτό δεν είναι εύκολο, έπρεπε να διαπραγματευτούν ε, με τις αποσχιστικές αρχές. Επίσης υπάρχει κίνδυνος οι αρχές να τους επιτρέψουν να δουν μόνο αυτά που θέλουν να δείξουν, για να μας αναφέρουν μόνο αυτά που, θέλουμε, που θέλουν να ακούσουμε να κίνδυνος βέβαια από τον οποίο γνωρίζουμε. Έχουμε εξοπλισμό για να παρακολουθούμε από αέρος την κατάσταση, δηλαδή έχουμε μη επανδρομένα υπτάμενα οχήματα, Δηλαδή, διαρκώς συναντούν σοβαρά εμπόδια και σε καμία περίπτωση καταρρίφθηκαν με αντιεροπορικά πυρά. Ε, άλλες φορές υπήρξαν ε, παράσιτα στα συστήματα επικοινωνίας. Μπήκαν δηλαδή στις, στις ε, που είχαμε εμείς για αυτή την επιχείρηση και μάλιστα οι δικοί μας μας είπαν ότι ήταν πολύ υψηλή τεχνολογία, στρατιωτική καπαράσιτα. Τώρα έχουμε εμείς πάρει μέτρα για να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο και να μπορέσουμε και πάλι να λειτουργήσουμε. Τώρα, η εντολή παρακολούθησης και παρατήρησης έχει εξελιχθεί και μετατραπεί σε επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης. Μιλάμε για πάυση του πυρό, αλλά η πάυση του πυρός δεν υπάρχει. Έχουμε σοβαρές ανησυχίες ασφάλειας για το προσωπικό μας που είναι όλοι ε, άοπλοι πολίτες ε, και γι' αυτό και δεν πρέπει να του εκθέτουμε σε κίνδυνο. Αυτό είναι ένας πρακτικός περιορισμός που ε, περιορίζει την ελευθερία κινήσεών μας. Επίση θέλουμε να αποφύγουμε μια κατάσταση όπου έχουμε πρόσβαση μόνο μέχρι τη γραμμή πάυσης των εχθροπραξιών ή εν πάση τη γραμμή των εχθροπραξιών, όπως θέλετε πείτε τι, για να μην τραβάμε γραμμές επί του εδάφους. Δηλαδή από το μέτωπο μέχρι το, τα σύνορα, ε, γιατί τα σύνορα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Αναφέρεται αυτό και στη Συμφωνία του Μίσκ και πάλι να σας πω ότι δεν έχουμε πρόσβαση μέχρι τα σύνορα. Το μόνο άμεσο σημείο που, ε, παρατήρησης που έχουμε όσον αφορά τη διέλευση των συνόρων είναι μια συμφωνία με τη Ρωσική Ομοσπονδία που έχουμε μια επιχείρηση στα ρωσικά σύνορα σε δύο φυλάκια όπου έχουμε την εντολή να παρακολουθούμε, να παρατηρούμε την διέλευση και είδαμε ρωσικά δίθεν ανθρωπιστικά ε, κομβόη, δεν τα επιθεωρήσαμε και αυτό το κάναμε στην συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό γιατί προσπαθούμε να, τους να το αντιμετωπίσουμε ως ανθρωπιστική επιχείρηση. Ο Ερυθρός Σταυρός δεν βρήκε συμφωνία ούτε με τους Ρώσους ούτε με τους ε, αποσχιστές ε, που όσον αφορά την διανομή της βοήθειας, εμείς μείναμε δηλαδή εκτός και παρατηρήσαμε απλώς το πέρασμα των φορτηγών και τώρα είναι στο δρόμο κι άλλο ένα κομβόι. Όσον αφορά τώρα τη συνεννόηση, ε, νέοι μηχανισμοί φάνηκαν επί τόπου. Ε, η Κοινή Επιτροπή, όπως λέγεται, Joint Commission, CCC, που όμως μέχρι στιγμή δεν έχει δείξει μεγάλες ε, ικανότητες να ασκήσει έλεγχο, της έλεγχο της κατάστασης. Πρόκειται για μια επιτροπή όπου οι Ρώσοι στρατικοί εκπρόσωποι ε, συνεδριάζουν με τους Ουκρανούς αλλά και με τους εκπροσώπους των αποσυστικών ε, ομάδων. Ε, Εμεί παρακολουθούμε μόνο, παρατηρητές είμαστε. Αν δούμε ότι μπορεί και να υπάρξει κάποια δυνατότητα αποκλιμάκωσης, θα εμπλακούμε πιο άμεσα, αλλά για την ώρα θεωρούμε πως είναι περισσότερο μία κίνηση, περισσότερο εντυπωσιασμού γιατί, και γι' αυτό και κρατάμε μια απόσταση γιατί μπορεί έτσι να νομιμοποιήσουμε και τους εκπροσώπους αυτών των ομάδων να ενισχύσουμε δηλαδή το στάτους τους γιατί γίνανε και τοπικές εκλογές πρόσφατα όπου φυσικά εμείς δεν τις αναγνωρίζουμε τις ε, θεωρούμε παράνομες γιατί δεν αντιπροσωπεύουν, δεν, δεν αντιπροσωπεύουν την υγρονική νομοθεσία. Συνεργασία με την Ένωση είναι υποστήριξη γιατί ε, ε, το 70% προέρχεται από τις χώρες της Ένωσης, ε, εξαιρετικά ισχυρή δηλαδή συμβολή και για την οποία είμαστε πολύ ευγνώμονες. Βέβαια, ο ΑΣΕ δεσμεύεται σε διάφορα θέματα όπως η παρατήρηση εκλογών, μεγαλύτερη μας επιχείρηση για τις προεδρικές και τις κοινοβουλευτικές ε, εκλογές ήταν στην Ουκρανία και ακούω και οι σχέσεις με το Ευρωκοινοβούλιο ήταν πολύ καλές, οπότε πρόκειται για έναν τομέα όπου νομίζω είμαστε ευθυγραμμισμένοι και κάνουμε το σωστό μαζί. Όμως αν δούμε την ευρύτερη εικόνα, ε, θα πρέπει να ανησυχούμε. Για την Ουκρανία η πολιτική διαδικουσία δεν έχει προχωρήσει όσο θα έπρεπε. Βλέπουμε κάποιες εξελίξεις οι οποίες μας φαίνονται ανησυχητικές. Προσπαθώντας να διευρύνουμε τώρα την εικόνα μας βλέπουμε ότι υπάρχουν ανησυχητικές εξελίξεις και στην Γεωργία. Βλέπουμε τις συμφωνίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Απχαζία οδηγούν σε μια στενή μορφή συνεργασίας για την ενσωμάτωση και την ασφάλεια της Αυγαζίας με τα σύνορα ανάμεσα στις δύο περιοχές να εξαφανίζονται ουσιαστικά και η Ρωσία να αποκτά νέα σύνορα με την Γεωργία και το ίδιο φαίνεται ότι γίνεται και στην Οσετία. Στην υπερνηστερία οι διαπραγματεύσεις δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Οι τελευταίες συναντήσεις του 5 όπου εκπροσωπείται και η Ένωση, ακυρώθηκαν. Τώρα γίνονται εκλογές και δεν υπάρχουν προοπτικές για την επανέναρξη της διαδικασίας. Και υπάρχει και το θέμα της γκαγκαουζίας και υπάρχουν και ερωτηματικά για τις εκλογές φυσικά. Ο Υπουργός ή Υπουργός ή Πρωθυπουργός της Μολδαβίας μου είπε ότι η μαζική προπαγάνδα την οποία βλέπει στα κανάλια που ελέγχονται από τη Ρωσία είναι κάτι το πολύ ανησυχητικό και είναι αντίστοιχο με αυτά τα οποία βλέπουμε στην Ανατολική Ουκρανία όπου υπάρχει ένας πραγματικός πόλεμος ενημέρωσης και κάποια κανάλια κλείνουν, αντικαθίστανται οι κεραίες, και γενικά ο αγώνας ανάμεσα στις δύο πλευρές σε επίπεδο μέσων ενημέρωσης είναι πάρα πολύ πολλωμένος. Όπως ήμουνα εκτός άκουσα ότι οι Αζέρι κατέριψαν ένα αρμενικό ελικόπτερο και υπάρχουν θύματα και μας ανησυχεί αυτό ε, γύρω από το Άνω Καραμπάχ, το πώς εξελίσσεται η κατάσταση και τέτοιου είδους συμβάντα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σαν σπινθήρας κρίσης σε μια περιοχή η οποία είναι από τη φύση της ασταθής. Το ίδιο ισχύει και στην Κεντρική Ασία. Υπάρχει μια κάποια ε, κατάσταση εκνευρισμού ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται η κρίση δημιουργεί ρηγματα στις κοινωνίες. Έχουμε μεγάλες ρωσόφωνες κοινότητες στις χώρες αυτές, οι οποίες έχουν έρθει σε επαφή μεταξύ τους με τα χρόνια και τώρα φαίνεται ότι υπολώνεται η κατάσταση επίσης και σε θρησκευτικό επίπεδο που θα μπορούσε να επηρεάσει τις χώρες της περιοχής. Ζητώ συγγνώμη για την ταχύτητα με την οποία παρουσιάζω όλα αυτά τα θέματα, αλλά η κατάσταση είναι προβληματική. Και ακριβώς γι' αυτό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία εγώ θεωρώ σαν βασικό θεμέλιο της ΟΑΣΕ, πρέπει να υπάρξει μια ισχυρότερη εμπλοκή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να ευνοεί, να είναι πιο καθοριστική η παρέμβασή σας για την αποφυγή εν πάση περιπτώσει σειράξεων, για την επιβολή κυρώσεων, αλλά απαιτείται ταυτόχρονα να συνεχιστεί και η πολιτική η οποία έχει σαν στόχο την επαφή και τις προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων. Και άλλωστε ο χώρος τον οποίο εκπροσωπώ, ο ΑΣΕ, αυτό έχει σαν βασικό στόχο. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να επιβάλλουμε ακριβώς αυτή τη λογική, τη λεγόμενη Ελσίνκη συν 4, ε, ένα κομμάτι δηλαδή της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μέχρι τώρα η συμμετοχή της Ρωσίας ήταν σχετικά περιορισμένη. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη βλέπουμε ότι παραβιάζονται βασικές αρχές της οργάνωσης και του διεθνούς συνταγματικού δικαίου από πλευράς της Ρωσίας, κάτι το οποίο καθορίζει τις σχέσεις μας τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια. Το ότι υπάρχουν όμως αυτές οι παραβιάσεις δεν πρέπει να μας αποτρέψει από το να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε τα θέματα. Ακούμε από πλευρά Ρωσία ότι αυτό που λέμε εμεί παραβιάσεις δεν είναι παραβιάσεις αλλά ότι οι κανόνε του παιχνιδιού δεν αντιστοιχούν με τι δικές τους ανάγκε και τα δικά τους χαρακτηριστικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο δίδει κάποιε εξηγήσει για την πορεία που έχει η κατάσταση και την έλλειψη σταθερότητα. Στη Βασιλεία προβλέπεται το Δεκέμβριο συνάντηση υπουργών του ΟΑΣΕ υπό την Προεδρία των Σέρβων αυτή τη φορά ακολουθεί μια υποψηφιότητα γερμανικής προεδρίας, ελπίζω να, είναι, να γίνει δεκτή και είναι καλό για την οργάνωση ε, να υπάρχει ένας ισχυρός υπουργός, μια ισχυρή χώρα. Η Σερβία προσπαθεί να λειτουργήσει σαν ειλικρινής ενδιάμεσος ανάμεσα στην Δύση και την Ρωσία. Ε, Θέλουν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση οι Σέρβοι και θέλουν ε, να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους χρησιμοποιήσει για να έχει καλύτερες επαφές με τον ρωσικό παράγοντα. Λοιπόν, αυτά. Φοβάμαι ότι δεν έχω πάρα πολύ χρόνο πλέον στη διάθεσή μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Ίσως μια-δυο ερωτήσεις, αλλά πρέπει να πάμε στην Ολομέλη έτσι κι αλλιώς. Έχετε πληροφορίες για μετακίνηση στρατευμάτων όχι μόνο στο Λούγκανς και στο Ντόνσκα αλλά και στο Μπραζέτους και αλλού γύρω από την Μαριούπολη. Και από την Κρυμαία προς την Οδέσα. υπάρχει καμιά τέτοια πληροφορία για τέτοιες προετοιμασίες. Εμείς μπορούμε να πούμε για αυτά που βλέπουμε. Για την Μαριούπολη δύο πράγματα. Η Μαριούπολη είναι εκεί που στείλαμε εμεί ένα από τα μη επανδρομένα σκάφη μας που χτυπήθηκε. Κάποιος δηλαδή μας εμπόδισε να το κάνουμε. Κάτι σημαίνει αυτό. Δεύτερον, η Μαριούπολη εξακολουθεί να είναι από τις περιοχές που έχουν μεγάλο πυροβιλικό. Από την πλευρά των αυτονομιστών, ναι. Άρα και αυτό θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι προετοιμασία για στρατιωτική παρέμβαση. Αυτά είναι τα πράγματα που βλέπουμε, αλλά δεν έχουμε πρόσβαση από εκεί και πέρα. Όταν συζητάμε με τους Ρώσους για την εφαρμογή συμφωνιών, είναι πολύ σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση να λέμε στους Ρώσους ότι και αυτοί πρέπει να προσπαθήσουν να διευκολύνουν την πρόσβαση στους διεθνείς παρατηρητές. Αλλιώς δημιουργούν υπόνοιες για κακή πίστη όσον αφορά την εφαρμογή των συμφωνιών. Ωραία, ερωτήσεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια σύντομη ερώτηση. Σήμερα διάβασα ότι ίσως οι Ρώσοι ήδη στην Κρυμαία έχουν κάποιες πυρηνικές δυνατότητες ή εν πάση περιπτώσει δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών μονάδων. Εσείς μπορείτε να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό, είναι αλήθεια, ισχύει. Όχι. Το ΝΑΤΟ έχει βέβαια δορυφορικές εικόνες, εμείς όχι, δεν ξέρουμε. Εμείς χρησιμοποιούμε μόνο ό,τι έχει ήδη συμφωνηθεί. Στην Κρυμαία δεν έχουμε πρόσβαση. Είχαμε στην Σεβαστούπολη και η Ουκρανία θέλει να το κλείσει. Δυστυχώς δεν μπορούμε εξαιτία της Ουκρανίας να πάμε εκεί. Η εντολή της υπηρεσίας καλύπτει την Κρυμαία, αλλά δεν έχουμε πρόσβαση εκεί. Που είναι πρόβλημα και γενικότερα για τους τάρταρους στη μειονότητα εκεί. Δεν μπορούμε να πάμε και να τους προστατεύσουμε. Για τα πυρηνικά δεν έχω καμία πληροφορία. Αμφιβάλλω να πρόκειται για πηγή όσα τα ΟΑΣΕ τα μέσα ενημέρωση φυσικά γράφουν διάφορα, αλλά από τον ΟΑΣΕ δεν νομίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο. Ωραία, την επόμενη φορά θα έχουμε περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε και τη σχέση μας και με τον ΟΑΣΕΦ. Σας ευχαριστούμε πολύ.